γυναίκες, ε, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα επίσης πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Και βεβαίως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα θέματα υγείας ε, και ασφαλείας για να υπάρχει και ο πλανήτης και στο μέλλον. Όλα αυτά πρέπει να γίνει για να έχουμε μια πιο δίκαιη συνεργασία να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις αυτές ε, και να πολεμήσουμε τη φτώχεια και την ανισότητα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Άλεξ Άγγιου Σαλίμπα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχει αλλάξει σημαντικά ο κόσμος μετά τη συμφωνία του Κορτονού και την έγκρισή της πριν από 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν σε μια νέα εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ ε, οι διπραγματεύσεις μας πρέπει να οδηγήσουν σε μια φιλόδοξη και σφαιρική ε, πολιτική συνένεση που θα οδηγήσει ε, στη μια βιώσιμη ανάπτυξη συμπεριληπτική και θα επικεντρώνεται σε ζητήματα πολύ σημαντικά όπως δημοκρατικά, ανθρώπινα δικαιώματα, οικονομική ανάπτυξη και απέντηση, κλιματική αλλαγή, εκρίζωση τη φτώχεια, ειρήνη και ασφάλεια, μετανάστευση και κινητικότητα. Επιπλέον, θα ήθελα να, ήθελα να υπογραμμίσουμε τη σημασία του να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση τη μελλοντική συμφωνία που πρέπει να εξασφαλίζει δημοκρατική λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα. Είναι κεφαλαιόδες λοιπόν η Ευρωπαϊκή η, η κοινή κοινοβουλευτική ε, επιτροπή ε, ΑΚΕ, και Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει να συνεδριάζει δύο φορέ το χρόνο σε ολομέλεια και μια φορά το χρόνο σε κάθε μία από τις τρεις περιοχές. Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμες, κρίσιμοι, μιας και μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στις σχέσεις μας με τις χώρες ΑΚΕ. Αυτό είναι κάτι που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη ε, της σχέσης μας ήπειρο προς ήπειρο με την Αφρική. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Τζούλη Βόρτ για ένα λεπτό. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών ΑΚΕ, γνωστή ω Συμφωνία του Κοτονού, ε, υπογράφηκε το 2000 και ολοκληρώνεται το 2020. Οι πραγματεύσει ε, για την διάδοχη κατάσταση είναι να εξελίξει και πρέπει να μην ξεχνάμε γιατί είναι σημαντική αυτή η εταιρική σχέση. Έχει αναπτύξει ένα πολιτικό διάλογο πολύ σημαντικό. Έχει αναπτύξει τη σχέση μεταξύ ημών και των χωρών και μέσω ενό πλαισίου που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Έχει επιτρέψει σημαντικέ συζητήσει να λάβουν χώρα για ζητήματα όπω η ελευθερία, ε, οι διακρίσει, ε, ε, σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική ταυτότητα, την σεξουαλική και αναπαρογική εκπαίδευση, καθώς και την ε, ε, εταιρική ευθύνη και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Πρέπει να ενισχύσουμε το χώρο, την, την, την εργασία στις χώρες και πρέπει να δώσουμε έμφαση στην κοινοβουλευτική διάσταση της Συμμετοχικής Συμφωνίας και να εξασφαλίσουμε δημοκρατική λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα και να προωθήσουμε ε, την ορατότητα και την αξιοπιστία αυτής της ε, ε, συμφωνίας. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και θα βασίζεται στην ατζέντα 2020 με μηχανισμούς αξιολόγησης ομοτήμων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους. Θα μπορούμε να έχουμε από κοινού μια, μεγάλη, μια πολύ ηχηρή φωνή παγκοσμίω να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις και πρέπει αυτό να το αποκαταπτρίσει και η συμφωνία. Σας ευχαριστούμε. Στα πλαίσια του Catch the Eye έχω λάβει δύο αιτήματα. Πρώτος θα μιλήσει ο κύριος Χουαν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Μίμητσα, σας χαιρετίζω ε, και αναγνωρίζω πολύ σημαντικό ρόλο σας τελευταία αυτή συνεδρίαση, μιας και ε, εδώ μιλάμε για τη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και με τι χώρε του 78 χώρε, μια συμφωνία που λύγει μετά από 20 χρόνια. Θέλουμε να ενισχύσουμε ε, την ρόλο των ε, τη κοινωνία των πολιτών και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πρέπει να παραμείνει ζωντανή αυτή η ε, κοινοβουλευτική διπλωματία. Είναι ένας, ένα εργαλείο οριζόντιου διαλόγου και αυτό δείχνει το γιγάντιο, γιγάντια προσπάθεια που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη, στην ευρωπαϊκή βοήθεια, ε, πάντα με βάση τι αξίε μα. Δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο τη πολιτική επιστροφών ή του ελέγχου τη μετανάστευση. Θέλουμε να, να ανταλλάξουμε εμπειρίες ε, στον τομέα της ε, ε, ενίσχυση του Κράτου δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ένταξης, τη καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και βεβαίω για να μπορέσει ο ρόλο των γυναικών να γιγαντωθεί στις χώρες της Αφρικής και τη Καραβική και του Ειρηνικού. Η Αφρική βεβαίω είναι ο γίγαντα εδώ. Η Αφρική είναι ο βασικό συνομιλητή τη Ένωση. Πραγματικά ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη κυρία Βοντελάιν που ψηφίστηκε σήμερα να φέρει σε πέρα αυτή τη διαπραγμάτευση και να μην ξεχνάει το ρόλο του, ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτήν την συμφωνία. Σα ευχαριστώ. Η Ρένα Γιώβεν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραβρέθηκα κι εγώ εκεί και είδα πραγματικά το τι σημαίνει αυτή η συνεργασία. Οι χώρε σε διάφορε υπήρου μπορεί να βελτιώσουν τι συνθήκε, ε, την ισότητα, την ειρήνη, ε, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και τα λοιπά. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα έγγραφο το οποίο θα επηρεάσει τη μελλοντική συνεργασία με τις χώρες ε, ΑΚΕ. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ευρωβουλευτές να παίξουν τον ρόλο τους στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Τώρα θα αναβαθμίσουμε την υφιστάμενη συμφωνία και το ψήφισμα αυτό βεβαίως ε, αναφέρεται και στον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Μαζί λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια επιτυχημένη κοινωνία και επιτυχημένες χώρες. Σας ευχαριστώ. Και τώρα εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο έχει πάλι και ο επίτροπο Νέβεν Μίμητσα. Παρακαλώ κύριε Επιτροπέ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Υπουργέ. Από την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, στις 28 Σεπτεμβρίου του 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες ε, ΑΚΕ έχουν διανύσει σημαντικό δρόμο κατά την προσπάθεια φυριλά μελλοντικής μας εταιρικής σχέσης. Και μάλιστα για μένα ήταν τιμή και προνόμιο και μεγάλη πρόκληση ότι ήμουν επικεφαλή τη διαπραγματεύτική ομάδα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι σε λίγο σχετικά χρονικό διάστημα επιτελέσαμε αισθητή πρόοδο. Η Γιούτα Αρπιλάινεν, ε, διάδοχός μου, θα έχει μια στέρεη και σφαιρική βάση ώστε να φέρει αίσιο πέρα στι διαπραγματεύσει. Είμαι αισιόδοξο ότι κάποια σημεία των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται ε, αυτή τη στιγμή σε παρενθέσεις που αντανακλούν κάποιες διαφορές μας και κάποιες εκκρεμότητες που έχουν μείνει και σημεία που θα πρέπει να συζητηθούν στο μέλλον δεν ε, είναι πουδενή ανυπέρβλητα εμπόδια που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την τελική συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο της μελλοντική συμφωνίας με τις χώρες και μετά το Κοτονού. Αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία θέλει κάποιο χρόνο φυσικά για να ολοκληρωθεί. Είναι περισσότερο θέμα χρόνου παρά έλλειψης πολιτικής βούλησης των συμβαλωμένων μερών η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η υποστήριξη και η ε, ανάμειξη, ενεργός ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση της συμφωνίας. Και θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμείνει στην προάσπιση των αρχών και αξιών της κατά την εταιρική της σχέση με κατά την εταιρική της σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Και τώρα εκ μέρους του Συμβουλίου το λόγο έχει η κυρία Τίτη Τουπουράινεν. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, Τα θέματα μετά το Κοτονού είναι πολύ βασικό θέμα για το Συμβούλιο. Σας διαβεβαιώ. Δράτουμε επίσης ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Επίτροπο τον κύριο Νίμιτσα για την ε, δουλειά που έχει κάνει. Εφαρμόζουμε λοιπόν την ατζέντα του 30 και τη Συμφωνία των ε, Παρισίων και βεβαίως για να αλλάξουμε το... και έχουμε και το παγκόσμιο πλαίσιο το οποίο αλλάζει, τις νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες. Πιστεύουμε ότι η ατζέντα του 2030 και η Συμφωνία των ε, Παρισίων ε, θα πρέπει να διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας και στα πιο δύσκολα ζητήματα. Ως Φιλανδική Προεδρία αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις διαπραγματεύσεις και θα προσπαθήσουμε το Συμβούλιο να συνεισφέρει στην πρόοδο αυτού του θέματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι για τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Έχω λάβει ένα σχέδιο ψηφίσματος κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης. Η ψηφοφορία του θα γίνει αύριο. Συνεχίζουμε αύριο στις 28 ε, Νοεμβρίου. 2019 από 9 μέχρι 12.30 και από 3 μέχρι 4. Και μάλιστα έχουμε τις σχετικές δημοσίευσεις στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλό βράδυ.